Κυρίες και κύριοι, ε, τα πρακτικά έχουν διανεμηθεί. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασής μας. Το Συμβούλιο διαβίβασε στο Κοινοβούλιο